λοιπόν Θα υποβάλλουμε για έγκριση τα πρακτικά πριν την επόμενη σύνοδο. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσει, τα ψηφίσματα τα οποία εγκρίθηκαν θα διαβιβαστούν στα αρμόδια ε, σώματα τα οποία αναφέρονται στη συγκεκριμένη ε, στον κύριο ψήφισμα. Σας εύχομαι καλή επιστροφή. Σας ευχαριστώ για τη συνεργασία και το ίδιο ισχύει και για του.